Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας που είναι ολοήμερη και λέγεται Περιφερειακή Επιτροπή. Το επόμενο θέμα είναι ψηφοφορία. Μία έκθεση. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Κοντ, ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Αριμόντ υπέβαλε τη σχέδιο γνωμοδότησής του στις 4 Νοεμβρίου και η, κατάθεση, η διορία για την κατάθεση των προϊόντων έλξη στις 13 Νοεμβρίου. 48 τροπολογίες κατατέθηκαν και μερικές συμβιβαστικές επετεύχθησαν. Πριν περάσουμε όμως την ψηφοφορία, μήπως ο εισηγητής κύριος Αριμόντ θέλει να μας πει τίποτε. Όχι, όχι, όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, Λέτε να κάνουμε κανέναν έλεγχο. Καλά. Με ποιο ερώτημα, ποιο θέμα. Έλεγχος των μηχανημάτων. Έλεγχος των μηχανημάτων άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Κύριε εντάξει, δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει. Παντού, παντού, παντού. Δεν είδατε το αποτέλεσμα. Α. Λοιπόν, ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα δουλεύει λέει. Έληξε η ψηφοφορία. Μάλιστα. Τώρα δουλεύει. Δουλεύει. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στο τέλος της εξέτασης των τροπολογιών. Τα υπόλοιπα διανοτάσεως της χειρός. Παράγραφος ένα νέα. Νέα συμβιβαστική υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Πόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απαρρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές απαρρίπτεται. Συμβιβαστική τρία. υπέρ κατά αποχές No objection. Α, ναι, απορρίπτεται. Όχι. Εγκρίνεται Εννέα υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται συμβιβαστική τέσσερα υπέρ κατά χές εγκρίνεται Συμβιβαστική 5 υπέρ. Υπέρ ξανά. Κατά. Εσ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. 6. 6 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές παρήπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 σε τμήματα σε τέσσερα τμήματα. Τέσσερα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. υπέρ Κατά. Χες. Γίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Τροφολογία 31. Υπέρ κατά που ρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές παρίπτεται 33 υπέρ κατά παρίπτεται Απαρρίπτεται. 40 υπέρ κατά χες παρρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αρχές επαλήθευση για την 43 παρακαλώ ηλεκτρονικός Α, δεν δουλεύοντας ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ευχαριστώ. Έληξε. Απαρρίπτεται. Απαρρίπτεται. 46 υπέρ κατά εποχές παρύπτεται. Τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Α, όχι, όχι γνωμοδότηση. Είναι η σφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το 2004 το Συμβούλιο ενέκρινε μία απόφαση για το τωρινό άρθρο 349 της Συνθήκης που έδινε το δικαίωμα στη Γαλλία να εφαρμόζει δεκαετή περίοδο εξαίρεση από τις μειώσεις του Dog Tax για τις γαλλικές απόκεντρες περιοχές. Και το Συμβούλιο μετά ζήτησε να παραταθεί το καθεστώς αυτό και να δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 15 <coughs> μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου 20. Η πρόταση αυτή εξετάζεται με την διαδικασία διαβούλευση στο Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά μόνον αφού έχει ακουστεί η άποψη του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η διαβούλευση. Η Κομισιόν ενέκρινε την πρότασή της πολύ αργά για μας, ώστε να την εξετάσουμε στη συνεδρίασή μας των αρχών Νοεμβρίου. Και αυτό έθεσε το Κοινοβούλιο σε πολλή πίεση, γιατί αν δεν εγκριθεί πριν το τέλος του χρόνου, τότε ο νέος νόμος, τότε ο παλαιός θα συνεχίσει να ισχύει και θα, θα καταργηθεί μάλλον και θα υπάρξει νομικό κενό. Αυτά κάνουν οι καθυστερήσεις και θα το θέσω και με τη νέα Επιτροπή αυτό το θέμα. Στο μέλλον η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίζει ότι θα προσαρμόζει, θα, επιβάλλει, θα υποβάλει τις προτάσεις της ΕΝΚΕΡ στο Κοινοβούλιο για να μην χρειάζεται πίεση. Και είναι κατεπίγουσα, οι συντονιστές συμφώνησαν, η πρόεδρος, να γράψει μία εκθεσούλα υπό την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 15. Υπό τη διαδικασία αυτή η πρόεδρος μπορεί να προτείνει μια, να εγκριθεί μία νομοθετική πρόταση χωρίς τροπολογίες εκτός εάν ένα δέκατο των μελών της Επιτροπής αντιτίθεται. Και τότε γράφει έκθεση στην Ολομέλεια η πρόεδρος το Δεκέμβριο εγκρίνοντας την πρόταση. Μετά την εξήγηση αυτή λοιπόν. Μπορώ να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν αντιρρήσεις. Έχουν. Δεν έχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την, ολομέλεια, την έκθεση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Εκ καρδίας. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Έχετε τις αποφάσεις. They were sent at Απεστάλησαν κατά τις 2 το μεσημέρι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στις αποφάσεις αυτές Λέει η πρόεδρος και διακόπτη. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ε, την υποβολή επίσημης έκθεσης από την κυρία Κρέτσου. Στην κυρία Κρέτσου. Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή, αλλά η επίσημη έκθεση θα χρειαστεί πολύ χρόνο μέχρι να συνταχθεί. Με αυτές τις αλλαγές εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο έγγραφο. No. Okay. Thank you. Thank you. And our next point. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης Είναι και το βασικότερο του απογεύματος. Θα ήθελα να καλωσορίσω τρεις ανώτατους αξιωματούχους από τη Γενική Διεύθυνση Ρίγκιο για ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη νέα γενεά της πολιτικής συνοχής. Ο καθένας θα κάνει μια παρουσίαση 15 λεπτών για τους τομείς που, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Μετά θα προβούμε σε ένα γύρο ερωταποκρίσεων μετά από κάθε παρουσίαση και αυτή η ανταλλαγή, μάλλον η συνεδρίαση ερωταποκρίσεων θα κρατήσει 30 λεπτά όπως σας είπα σήμερα το πρωί. Ο κύριος Νίκολας Μάρτιν, αναπληρωτής υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της πολιτικής μας και θα μας μιλήσει για τον προγραμματισμό στη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Τιμή μου που είμαι εδώ και έχω την ευκαιρία να σας δώσω μια γενική εικόνα για το ποια είναι τα βασικά σημεία της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, του 2014 μέχρι 2020 βεβαίως θα παρουσιάσω το αποτέλεσμα μακροσκελών διαπραγματεύσεων το οποίο επετεύχθη χάρη και στην στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ πέρα πραγματικά οφείλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συμβολή του χάρη στην οποία τελικά καταλήξαμε σε μια νέα εξυγχρονισμένη πολιτική συνοχής. Ελπίζω λοιπόν mm η παρουσίαση υπεριμφερόταν σε Τι έγινε τώρα. Τέλος πάντων. ελπίζω να εμφανιστεί. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είμαι εδώ με δύο συναδέλφους διευθυντές το τη Γενική Διεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Πολιτικής θα καλύψουμε τα εξής θέματα, να σας δώσω τα γενικά στοιχεία και μετά θα πω κάποια πράγματα για τον προγραμματισμό που κάνουμε τώρα. Και θέλω να τονίσω κάποια από τα στοιχεία αυτής της διαδικασίας και να σας πω πού βρισκόμαστε. Και μετά ο Ρουντόλφ θα αναφερθεί στο βασικό σημείο του εξυγχρονισμού. Και ο Φρανκ θα αναφερθεί στο κομμάτι του διαχειριστικού ελέγχου. Και βέβαια μετά θα δούμε τη διαδικασία απαλλαγής 2007 με 2013. Οπότε, ποια είναι τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης. Ε, τι είναι το διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα στοχεύουμε τους πόρους στους βασικούς τομείς ανάπτυξης για να φροντίσουμε πως τα λεφτά θα πάνε στις περιοχές υψηλής προτεραιότητας για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένους τρόπους. Ένας άλλος τρόπος για να γίνει πιο αποτελεσματική η χρηματοδότηση είναι να έχουμε αποτελεσματικά προαπαιτούμενα Ε, συντονισμένη χρήση για να μην δουλεύουμε απομονωμένα. αλλά να συνδεόμαστε με τον προγραμματισμό. Μετά η σχέση με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τις διαδικασίες μεταρρύθμισης. Εδώ πέρα μιλάμε για την οικονομική διαχείριση. Μετά ενισχύουμε την διαβεβαίωση στο τμήμα του ελέγχου και μετά απλοποίηση. Για την οποία πάλι θα πω κάποια πράγματα. Έχουν αλλάξει λοιπόν αρκετά πράγματα εδώ πέρα για το 2014-2015 σε σχέση με την περίοδο 2017-2013. Γι' αυτό λέμε πως έχουμε μια νέα πολιτική για αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο. Μια γρήγορη μετά παρουσίαση, αν δείτε την αρχιτεκτονική του 2007-2013 μιλάμε για σύγκληση και εδαφική συνεργασία. Τώρα έχουμε δύο στόχους που αντικατέστησαν τους προηγούμενους. Έχουμε επενδύσεις για ανάπτυξη και δουλειές που αφορά τη χρηματοδότηση των κρατών μελών, εδαφική συνεργασία και μετά αν δούμε τη χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη έχουμε τρεις κατηγορίες περιφερειών, τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Αυτό που λέγαμε σύγκληση, μετά έχουμε τις πιο ανεπτυγμένες, αυτό που λέγαμε παλιά ανταγωνιστικότητας. Ε, αυτά βεβαίως είναι ε, με βάση το ΑΕΠ κάτω από το 75%, άνω από το 90% και μετά τη νέα κατηγορία, κάτι μεταξύ των δύο, για να φανεί η αλλαγή, μια μεταβατική δηλαδή κατηγορία περιφερειών που ωφελούνται από συγκεκριμένους όρους. Και μετά όσον αφορά τη χρηματοδότηση βλέπετε εδώ την κατανομή που σας δίνει το νούμερο 351 δισεκατομμύρια και το μεγάλο ποσό βεβαίως πάει στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αλλά θα σας στείλω και της διαφάνειας. Κάτι άλλο σημαντικό που αφορά την συντονισμένη χρήση είναι το να έχουμε κοινού κανόνες για τα πέντε ταμεία, όχι μόνο την πολιτική συνοχή. όχι αυτά τα οποία ξέρετε, ΕΤΠΑ, Ταμείο συνοχή και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και το Ταμείο ε, Ανάπτυξης της υπαίθρου και αλίας. Γιατί ο στόχος μας ήταν να έχουμε ακριβώ κάποιους κοινού κανόνες για τα πέντε ταμεία. Αυτό το οποίο λέμε ο κανονισμός των κοινών ε, διατάξεων. Και αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε ε, κάποιες απλοποιήσεις που θα αναφέρω σε λίγο. Ας δούμε τώρα τον προγραμματισμό, το τι κάνουμε τώρα. Οι κανονισμοί ευθύθηκαν το τέλος του 2013 και βεβαίως ε, τα βασικά μέρη των ε, κανονισμών ήταν αντικείμενο συμφωνίας ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στις αρχές του 2013 εσκεμένα δόθηκε βάρος στα στοιχεία εκείνα τα οποία θα επέτρεπαν να προχωρήσει ένας άτυπος διάλογος μεταξύ των κρατών μελών για να ξεκινήσει η ε, διαδικασία των προγραμμάτων. Επισήμως ξεκινήσαμε φέτος. Έχουμε συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου υπογράφηκαν και μετά έχουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα. Θα σας δώσω τα νούμερα σε λίγο να δείτε πού βρισκόμαστε. Οπότε, βλέπετε εδώ πώς έχουν τα πράγματα. 46 επιχειρησιακά προγράμματα έχουν εγκριθεί. Είμαστε στη φάση έντονης δραστηριότητας αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω κάποια ουσιαστικά νούμερα. Είναι πολύ δυναμική η κατάσταση. Είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα από ό,τι πριν από ένα μήνα. Φαίνεται ότι καθώς πάμε προς το τέλος του έτους ε, έχουν συγκεντρωθεί τα κράτη-μέλη και έτσι και εμείς προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και οπωσδήποτε πάνω από τα μισά προγράμματα είτε θα εγκριθούν είτε θα είναι έτοιμα προς έγκριση οπότε μπορεί να γίνει μεταφορά της ε, έγκρισης ε, πληρωμών για το επόμενο έτος αλλά ελπίζω να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Βλέπετε πως τρία κράτη-μέλη, Δανία, Λιθουανία και Λετωνία έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους. Ένα άλλο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αφορούσε την θεματική εστίαση. Το είπα αυτό στην αρχή. όπου έχουμε ακριβώς ε, τους ε, βασικούς τομείς προτεραιότητας για να υπάρχει αποτελεσματικότερη χρήση και αυτό έγινε μέσω ενός μενού 11 θεματικών στόχων έτσι ώστε κάθε ευρώ να συνδέεται με έναν από αυτούς τους θεματικούς στόχους και βλέπετε εδώ πέρα μπλοκ αυτών των στόχων που συνδέονται με τη στρατηγική του 2020 έξυπνη αηφόρος ε, λοιπά και βλέπετε εδώ πέρα τους τέσσερις πρώτους για τη χρήση του ΕΤΠΑ, έρευνα και καινοτομία, πληροφορική τηλεπικοινωνίες ε, και η οικονομία χαμηλού άνθρακα και βιώσιμη ε, ανάπτυξη, 80% στις ναι, ναι. Ε, ε, φτωχότερες ε, περιοχές, 15% ε, Αυτά τα ποσοστά είναι στον κανονισμό και κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού βεβαίως φροντίσαμε να συμμορφωθούμε. Και τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Και το γεγονός ότι μπορέσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ε, σημαίνει πως έχουμε μεγάλες διαφορές από το παρελθόν, αλλά με βάση τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης σας δίνουμε μια εικόνα τώρα το που θα πάνε ακριβώς τα λεφτά. Έχει σπάσει εδώ πέρα λοιπόν ένα θεματικό στόχο, βλέπετε την ανάλυση. Αν δείτε τα τέσσερα πρώτα, υπάρχει βάρος στο, του ΕΤΠΑ στους τομείς ναι. αυτούς και αυτό δείχνει πως η θεματική εστίαση λειτουργεί και πήγαν τα λεφτά εκεί πέρα που θέλαμε. Ενδιαφέρον επίσης είναι το θέμα το υπαριθμόν 7 η υποδομή δικτύου και αν συγκρίνεται αυτό το νούμερο με το νούμερο για το 2007-2013 βλέπουμε μια μεγάλη μείωση. Άρα μετατοπίζονται τα κονδύλια από εκεί που ήταν όπου δίναμε βάρος στις υποδομές προς ε, τις πιο έξυπνες ε, επενδύσεις. Επίσης, βλέπουμε την συνέργεια στην χρήση των ε, ταμείων, ώστε πραγματικά συνδυάζουμε τα κονδύλια. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εταιρικέ σχέσεις με στόχο να υπάρχει αυτό ακριβώς το κοινό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και υπάρχει η δυνατότητα προγραμμάτων σε πολλά ταμεία να συνδέεται το ΕΤΠΑ με το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά το οποίο εκμεταλλεύτηκαν 16 κράτη-μέλη και ε, έχουμε άρα αποτελεσματικότερη χρήση των ταμείων και κοιτάμε καλύτερα το πώς συνδέονται τα ταμεία με το κόσμο, τον ορίζοντα 2020 κτλ. Και βεβαίως υπάρχει ο οδηγός προς τους δικαιούχους ε, της Κομισιόν για να μπορούν αυτοί να καταλάβουν το τι γίνεται. Κάτι άλλο για την εδαφική πτυχή, μέρος και αυτό των διαπραγματεύσεων, υπήρχε προσπάθεια να ενισχυθεί η εδαφική διάσταση και ειδικά οι επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Μεγάλο κομμάτι του ΕΤΠΑ πηγαίνει ούτως ή άλλως σε αστικές περιοχές γιατί αν εστιάζει κανείς σε αυτούς τους βασικούς τομείς τότε ε, προφανώς εκεί πέρα θα είναι και οι επιχειρήσεις. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης ε, και υπάρχει μια εγγύηση σε αρχές για ένα ελάχιστο ποσοστό των κονδυλίων από το ΕΤΠΑ. Και βλέπουμε πραγματικά πως τα κράτη-μέλη δίνουν τις, ε, την δυνατότητα και στη, τη χρηματοδότηση στις τοπικές αρχές. Και με τις καινοτόμες αυτές τις δράσεις θα υποστηρίξουμε αυτή την εστίαση στην αστική διάσταση. Οι άλλες ε, πτυχές ανέφερα σύντομα την, τις ολοκληρωμένες ε, δαφικές επενδύσεις, ε, εστιάζεται δηλαδή η χρηματοδότηση για να υπάρχει μια στρατηγική εδαφική προσέγγιση 21 κράτη-μέλη και βεβαίως υπάρχει η Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης ε, που μπήκε πλέον σε όλα τα ταμεία και θα τη χρησιμοποιήσουν 16 κράτη-μέλη. Οπότε βλέπετε πως ξεκινήσαμε νέους τρόπους σκέψης για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Μετά έχουμε προαπαιτούμενα ex ante. Ένας καινούριο μηχανισμός έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως υπάρχουν τα προαπαιτούμενα, υπάρχει το σωστό περιβάλλον. Το σκεπτικό είναι πως δεν έχει νόημα να ξοδεύουμε λεφτά σε μια περιοχή επενδύσεων όπου είτε δεν ε, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες είτε δεν υπάρχει μια σαφής στρατηγική για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση ή ε, δεν υπάρχουν οι σωστές εθνικές Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα προαπαιτούμενα εξ άντε, όπως η έξυπνη στρατηγική εξειδίκευση. Ε, μετά έχουμε την γενική απέτηση για μη διακριτική μεταχείριση της αναπηρίας, αλλά και των δημοσίων προμηθειών. Οπότε μπορούμε να ε, επιβεβαιώσουμε την συμμόρφωση και εδώ πέρα βλέπετε μια γενική εικόνα της αξιολόγησης. Το κόκκινο είναι εκεί όπου θεωρούμε πως ε, η θεματική η τα θεματικά προαπαιτούμενα εξ άντε ε, δεν εκπληρώνονται. Υπάρχουν πολλά κόκκινα βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι οπωσδήποτε αρνητικό γιατί σημαίνει πως ο μηχανισμός κάτι βρήκε. Αλλιώς θα στέλναμε λεφτά εκεί χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα προαπαιτούμενα. Οπότε το γεγονός ότι βρήκαμε όλες αυτές τις περιοχές όπου πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα είναι κατά την άποψή μου ένα θετικό μήνυμα και σημαίνει πως τώρα έχουμε σχέδια δράσης με τα κράτη-μέλη και θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν ε, τα σωστά αποτελέσματα μέχρι το 2016 μέχρι το τέλος του 2016 το θέμα τώρα της εταιρική σχέσης ήταν κρίσιμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχε αρκετά μεγάλη στήριξη. Και έτσι είχαμε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς, μια πράξη κατεξοδότηση που υιοθετήθηκε κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους και ήδη άρα υπήρχε στις ε, διαπραγματεύσεις καθώς καθόριζε τις ε, λεπτομέρειες ε, που έπρεπε να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για να υπάρχει αυτή η εταιρική σχέση, αλλά ισχύει σε ε, όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας εφαρμογής και θα παρακολουθούν πολύ στενά και θα αποτελέσει βέβαια στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Και η τελευταία μου διαφάνεια για την απλοποίηση, μια λέξη που τη ακούω όσο καιρό ασχολούμαι με την πολιτική συνοχής, ήταν κάτι το οποίο διέταχε την προετοιμασία του πακέτου μας και της διαπραγματεύσεις απλοποίηση για τους δικαιούχους, δηλαδή να μην ε, ε, εμποδίζεται κανείς επειδή είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα ταμεία. Τα είπαμε νομίζω τα περισσότερα, ηλεκτρονική συνοχή με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινή κανόνες σε όλα τα ταμεία για κάποιους τομείς όπως τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Και πάλι εδώ πέρα λοιπόν θα το ξαναδούμε αυτό όταν ολοκληρωθεί η ε, ανάλυση. Ποιες δηλαδή δυνατότητες εκμεταλλευθήκαμε και πώς μπορούμε να προωθήσουμε και να εμπνεύσουμε την περαιτέρω χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Θα σταματήσω εδώ για να δεχτώ και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Τώρα τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να, επιβάλλουν, ε, να υποβάλουν, με συγχωρείτε, ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μάρτιν, γιατί όπως ε, είπατε, Υπάρχει δυνατότητα καλύτερου συντονισμού μεταξύ ορίζοντα 2020 και της έρευνας που χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Από πλευράς Επιτροπής, από τον κύριο Κατάινεν, μέσα στα πλαίσια της Ήτρε, δεν έλαβα απάντηση, δηλαδή αν τα διαρθρωτικά ταμεία είναι αποκλειστικά για τις περιφέρειες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει συντονισμός. Τώρα είδατε τα επιχειρησιακά προγράμματα. Πώς μπορούμε να εργαστούμε τα επόμενα χρόνια κατά καλύτερο τρόπο ή κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό. Ένα συντονισμός δηλαδή όπως θα τον επιθυμούσαμε. Έτεριτς. Ευχαριστώ. Πολύ καλή παρουσίαση και άκρος ενδιαφέρουσα. Αν, ας βάλουμε ένα δυνητικό αν, υπάρχουν τα προαπαιτούμενα για μια περιφέρεια, υπάρχουν θέματα ε, κοινωνικού αποκλεισμού, κλιματικών αλλαγών και ελέγχου και ούτω καθεξής. Αρχίζει η χρηματοδότηση. Τι θα γίνει αν ε, με μία εκλογική διαδικασία αλλάξουν οι προτεραιότητες ε, του, της τοπικής κυβέρνησης. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, σε σχέση δηλαδή με την αρχική δέσμευση και υπογραφή και τις αλλαγές που επήλθαν μετά από τοπικές εκλογές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση η απόκληση, Άντερσον. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα ήθελα ένα αντίτυπο αυτής της παρουσίασης PowerPoint. Σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα είπατε ότι έχουν εγκριθεί 46 περίπου. Πόσο θα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν πριν αρχίσουν να ε, ισχύουν τα νέα προγράμματα. Και σε σχέση με αυτά που προαναφέρατε, δηλαδή εάν το ΕΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δοθούν πόροι σε ένα τομέα και αν στη συνέχεια γίνουν περικοπές, δηλαδή το μερίδιο αυτό του ΕΚΤ χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια των ε, ιδίων πόρων μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ιρλανδία οι υπεύθυνοι για την απασχόληση και την κατάρτιση είπαν θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μερίδιο για να καλύψουν το δικό τους προϋπολογισμό παρά να το ε, αποδώσουν σε αυτά τα project. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. κυρία Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την εξαιρετική παρουσίαση. Μία ερώτηση έχω για την προσέγγιση που αναφέρατε για τα νέα αυτά προγράμματα που βασίζονται στην τοπική ανάπτυξη. Μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και η συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών και νομίζω πως εδώ πέρα μπορεί να συνδυαστεί μια προσέγγιση top-down με άλλη μια bottom-up. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να λάβει μέρος η κοινωνία των πολιτών και στα άλλα προγράμματα, το ITI και τις καινοτόμες αστικές δράσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Μπρεσό. Και εγώ θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τη διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είπατε ότι ένα μέρος θα εγκριθεί και το άλλο θα εγκριθεί σε μία μεταγενέστερη φάση με βάση μία διαδικασία το όνομα της οποίας δεν θυμάμαι αλλά που θα ενταχθούν στο φετινό προϋπολογισμό, που εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσονται στο πολιετές. Εκεί όμως που χρειάζεται τροποποίηση με βάση το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί δεν υπάρχει πληρότητα ως προς την ε, τρέχουσα διαδικασία έγκρισης. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το εξής. Μόλις συμπληρωθεί η διαδικασία, η Επιτροπή θα εγκρίνει εκτός και αν υπάρχει μεταγενέστερη έγκριση μετά από αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που δεν μπορεί να γίνει πριν από τα μέσα του έτους, Μάιο-Ιούνιο, περίπου εκεί. Κάτι το οποίο για τις περιφέρειες σημαίνει ότι θα κινηθούν τον Οκτώβριο. Ας θεωρήσουμε ότι το Μάρτιο θα έχουμε ένα άλλο πακέτο περιφερειών για τις οποίες η έγκριση θα γίνει αμέσως μετά, εάν εγκριθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλάμε για μια συμφωνία με τη συμμετοχή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που επιτρέπει στα κράτη και τις περιφέρειες να αρχίσουν να εργαστούν προτρέχοντας ως προς τους πόρους. Ας θεωρήσουμε όμως ότι υπάρχει έγκριση και δεν θα υπάρξουν μεταγενέστερες ε, τροποποίησεις. Ίσως έτσι θα μπορούσε να υπάρξει μία επιτάχυνση γιατί πολλές ε, περιφέρειες θα χάσουν δύο χρόνια γιατί έχουν ήδη περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος έχετε βρει έναν τέτοιο τρόπο επιτάχυνσης έτσι ώστε να προκαταβληθούν τα χρήματα με ίδιους πόρους αλλά με ένα πλαίσιο εγγύησης. Άλλα ερωτήματα. Ο κύριος Λούερ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην θεωρηθεί επιφανειακό το θέμα που θα θίξω. Υπάρχουν ορισμένες ε, προαπαι... ορισμένα προαπαιτούμενα σε σχέση με τους παραλήπτες της χρηματοδότησης, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχέση με άλλες χώρες, ε, δηλαδή ε, αιτιολογήσεις ως προς την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. γιατί μπορεί να υπάρχει <laughs> δέσμευση με τις τοπικές αρχές για χρηματοδότηση. Μπορεί κανείς να συμπληρώνει φόρμες, να αρχίζει έναν διάλογο, αλλά ίσως να μην ξέρετε ότι έχει γίνει η χρηματοδότηση μέσω του ΕΤΠΑ ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα αρχίσω με την τελευταία. Ναι, πράγματι υπάρχουν προαπαιτούμενα για, την, για δημοσιοποίηση εάν ε, τύχεται χρηματοδότησης. Υπάρχουν στον κανονισμό και λεπτομεριακοί κανόνες Άρα όποιος είναι δικαιούχος χρηματοδότηση, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, θα πρέπει να ε, συμμορφωθεί με αυτά τα προαπαιτούμενα. Εάν πρόκειται για οδικό δίκτυο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έγινε χρηματοδότηση, θα πρέπει να εγγραφεί. Εάν ε, οργανώσετε ένα σεμινάριο θα πρέπει να υπάρχει στην τεκμηρίωση. Εάν δεν ε, πληρούνται αυτός ο όρος, ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα, γιατί δεν μπορείτε να τα λάβετε από τον ε, κοινοτικό προεπολισμό και να μην το αναφέρετε ρητά. Αυτό αποτελεί παραβίαση των κανόνων. Ως προς την ερώτηση της κυρίας Μπρεσό, γιατί μας απασχόλησε πραγματικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σε σχέση με αυτό το ζήτημα της ταχείας έγκρισης των προγραμμάτων 14-20. Όπως είπατε, υπάρχουν τρία σενάρια. Τα προγράμματα που εγκρίνονται πριν από το τέλος του έτους, μία σειρά προγραμμάτων που είναι έτοιμα προς έγκριση μέχρι το τέλος του έτους, αλλά δεν έχουμε χρόνο μέσα στα πλαίσια του κοινοτικού μηχανισμού να υπογράψουμε τα προγράμματα αυτά στην Επιτροπή. Και η τρίτη ομάδα είναι τα προγράμματα που δεν είναι έτοιμα προς έγκριση στο τέλος του χρόνου. Για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει διαδικασία μεταφοράς, δηλαδή όταν έχουν υπογραφεί αλλά δεν ε, έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Δηλαδή η Επιτροπή σε αυτήν την περίπτωση μεταφέρει τις πιστώσεις το Φεβρουάριο του 2015 και αρχίζουμε να εγκρίνουμε αυτά τα προγράμματα που ήταν σχεδόν έτοιμα τα τέλη Δεκεμβρίου. Για την τρίτη ομάδα, οι πιστώσεις υποχρεώσεων θα πρέπει να εγγραφούν εκ νέου στον ε, προπολογισμό στο 2015, στη χρήση 15. Αυτό σημαίνει αναθεώρηση του πολιετούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού περί πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό υπάρχει μεταφορά, γίνεται μεταφορά και η σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2015 έτσι ώστε να αυξηθεί το συνολικό ποσό των πιστώσεων ε, ανάληψης υποχρεώσεων. Η αναθεώρηση εγκρίνεται μέχρι την 1η Μαΐου, μπορεί να γίνει βεβαίως και γρηγορότερα, εάν ε, υπάρξει μια πιο γρήγορη διαδικασία και από πλευράς Επιτροπής θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εγκρίνουμε με σπουδή αυτό το πλαίσιο. εξορισμού αυτά τα προγράμματα δεν ήταν έτοιμα προς έγκριση στο τέλος του 2014. Έπρεπε να γίνει περισσότερη εργασία, από τα κράτη-μέλη να συζητήσουν με την Επιτροπή της Περαιτέρω Αλλαγές έτσι ώστε τα προγράμματα να είναι έτοιμα προς έγκριση και δεν ξέρουμε πάντα πότε θα γίνει αυτό. Ίσως το Φεβρουάριο, Μάρτιο ή Απρίλιο. Θα είναι έτοιμα αυτά τα υπόλοιπα προγράμματα και θα προβάλλουμε μία ταχεία διαδικασία έτσι ώστε να είναι έτοιμα και μόλις γίνει αναθεώρηση του πολιετούς θα μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε παρευθύς. Ως προς ε, μια διαδικασία αιρεσιμότητας για την έγκριση, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ε, υποαίρεση έγκρισης, αλλά οι πληρωμές μπορούν να επιλεγούν από την πρώτη Πρώτου 14. Άρα τα κράτη-μέλη ή οι περιφέρειες μπορούν να εργαστούν για τα σχέδια αυτά, τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη, έτσι ώστε να εγκριθούν με την Επιτροπή Εποπτεία και αναδρομικά να γίνει κάλυψη, να υπάρξει κάλυψη. Αυτό είναι δυνατόν και το κράτος μέλος γνωρίζει πότε ένα πρόγραμμα είναι έντιμο προς έγκριση. Άρα ο κίνδυνος είναι μικρότερος από πλευράς κράτους μέλους. Είμαστε πραγματιστές και σε επίπεδο μονάδας ε, εκτέλεσης είμαστε σε επαφή με τις αρχές του κράτους για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και κράτους. Άρα ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Ως προς την κοινωνία των πολιτών, η συμμετοχή της προβλέπεται μέσα στα πλαίσια του κώδικα συμπεριφοράς. Έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη των ε, τοπικών φορέων. Είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και νομίζω ότι οι ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές προωθούνται. Δηλαδή η αστική αρχή είναι επικεφαλής και μιλάμε για συμμετοχή σε κατώτερο επίπεδο από το περιφερειακό ή το εθνικό. Άρα η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει στην επεξεργασία της ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής μέσα στα πλαίσια της εταιρικής διαδικασίας και το ITI, δηλαδή η επένδυση, οι εδαφικές επενδύσεις σχετίζονται με τις περιφέρειες ή μικρότερες ενότητες. Αλλά όλα αυτά τα μέσα σχετίζονται με την εταιρική σχέση έτσι ώστε να υπάρχουν ε, περιθώρια για την κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσει το ρόλο της. Και αυτό θα το δούμε έμπρακτα. Νομίζω ότι κάλυψα τα προγράμματα, τα προσέγγιση προγράμματα και ελπίζω ότι όλα τα προγράμματα θα εγκριθούν μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους και εάν το σημείο εκκίνησης είναι η έγκριση του κανονισμού, τότε θα κινηθούμε και γρηγορότερα από το 13. Αυτό θα θέλαμε και εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο θέμα που θίξατε, γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για τη Βόρειο Ιρλανδία όλα τα προγράμματα του κοινωνικού ή περιφερειακού ταμείου θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον κανονισμό. Διαπραγματευόμαστε με το, το πρόγραμμα και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη ότι οι προτεραιότητες είναι σωστές για την χρηματοδότηση και υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σας ε, απαντήσω επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορούμε να τις δούμε διμερώς. Αλλά καλύτερα να το δείτε με τη σχετική γενική διένθεση. Ως προς το δυνητικό εάν, θεωρούμε ότι τα προγράμματά μας αποτελούν ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης. Πρόκειται για επταετή προγράμματα με τρία χρόνια εφαρμογής. Δεν πρόκειται για βραχυπρόθεσμα προγράμματα, αλλά για μία μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν πιστεύουμε να, ότι υπέρχουν αλλαγές κάθε έξι μήνες ή ένα χρόνο και οι προτεραιότητες ε, που συμφωνούνται μεταξύ περιφερειών, κρατών, ε, μελών και επιτροπής δεν έχουν σχέση με τις ε, τοπικές πολιτικές. Δηλαδή ορίζουμε προτεραιότητες που συμφωνούνται ευρέως. Οι εκλογικές αλλαγές δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει νέα προσέγγιση στο πρόγραμμα βεβαίως. Οι αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να προβάλλουν μια πρόταση τροποποίησης ενός προγράμματος αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Γιατί αλλάζουν οι συνθήκες, η αρχική ανάλυση δεδομένων δεν είναι τεκμηριωμένη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι απόλυτα λογικό και επιτρεπόμενο αλλά αυτό δεν έχει σχέση με, τον καλύτερο, με τις για τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρηματοδότησης και δαπάνης. Τέλος, συνέργειες. Πρόκειται και για το, πιο, για το πλέον δύσκολο ζήτημα εδώ. Ο νομοθέτης έχει εντάξει στον κανονισμό όλα τα στοιχεία για να τονιστούν οι συνέργειες το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μια κοινή προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ νωρίς ε, για να δούμε κατά πόσο το έχουμε επιτύχει, αλλά θέλουμε να το δούμε και μετά τον προγραμματισμό για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουν επέλθει αλλαγές σε σχέση ιδιαίτερα με τα χρήματα του ΕΤΠΑ για την έρευνα και την ε, καινοτομία, καθώς και τον ορίζοντα 2020. Δεν μπορώ να σας δώσω παραδείγματα επί του παρόντος, αλλά θα πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος και ελπίζω να μπορέσουμε να σας δώσουμε ε, μία απάντηση βάση στοιχείων στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ. Υποσχεθήκαμε ότι θα σας ρωτούσαμε συνέχεια. Αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Και θα σας ευχαριστήσω κύριε Μάρτιν για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρούντολφ Νέσλερ διευθυντή του τμήματος πολιτικής που θα μας μιλήσει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Έχουμε και τα, τις διαφάνειες. Έχετε λοιπόν και εσείς το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας περιγράψω το δεύτερο τμήμα της παρουσίασης που ασχολείται με το θέμα του πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής που ήταν ένα από τα κύρια θέματα που μας ενδιέφεραν και με οποία, για το οποίο μιλήσαμε και με σας όταν προγραμματίζαμε για πρώτη φορά την περίοδο. Θα τονίσω συγκεκριμένα θέματα που θέλω να θίξω. Το πρώτο είναι η αποτελεσματικότητα, το δεύτερο η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και τέλος θα σας πω μερικά πράγματα για τη χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων. To start with, uh, uh, it's Καταρχήν, πρέπει να τονίσουμε ότι στο παρελθόν η πολιτική συνοχής βασιζόταν κυρίως υπερβολικά στην δαπάνηση των πόρων της τούλες και λιγότερο με τα αποτελέσματά της. Στη νέα περίοδο, προγραμματική περίοδο συνεννοηθήκαμε με τα κράτη-μέλη και είπαμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς στόχο έχουμε. Τι στόχο. Θέλουμε να γνωρίζουμε καλά ποια είναι η λογική των παρεμβάσεών μας. Αυτό αφορά καταρχήν τι πρέπει να αλλάξει μέσω των παρεμβάσεων και των προτεραιοτήτων μας. Και γι' αυτό έχουμε μια κατηγορία δικτών που λέγονται «Result indicators Και επειδή το θέμα αφορά και τις δαπάνες, αυτούς τους πόρους τους διαθέτουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα βέβαια και θέλουμε να παρακολουθούμε και τι πρόοδος γίνεται ως προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε. Αυτό αφορά όπως καταλαβαίνετε το output. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο είδη δικτών και υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να τους χρησιμοποιούν τους δείκτες. Για να σας δείξω λιγάκι ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε εδώ το παράδειγμα που δείχνω. Γενικά αυτός ο δείκτης αποτελεσματικότητας σχετίζεται με τους στόχους του 2020, παραδείγματος χάρη, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας μιας περιφέρειας. Θέλουμε να, μετρήσουμε, να το μετρήσουμε αυτό μέσω της μείωσης του χρόνου που απαιτείται για να πάει κανείς να μεταβεί στην περιφέρεια αυτή ή για την αύξηση της, απο... της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που το μετράμε με την αξία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στα προγράμματά μας. Είναι αρκετά απλοί δείκτες και λογική Σύνδεσης αποτελέσματος με τον σχετικό του δείκτη. Πιο συγκεκριμένο ακόμα, για τους ε, δείκτες output. Εκεί μετράμε τι χρησιμοποιήσαμε πράγματι από τους πόρους μας. Αυτό παραδείγματο χάρη μπορεί να αφορά τον αριθμό επιχειρήσεων που στηρίχτηκαν ή τον αριθμό των ερευνητών που στηρίχτηκαν χιλιόμετρα δρόμου που δημιουργήθηκαν κλπ άμεσα αποτελέσματα δηλαδή που μπορούμε να έχουμε με τα δαβανηθέντα χαρήματα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο είδη δικτών και μεταξύ τους έχουμε και πολλούς υποχρεωτικούς. Διότι είναι σημαντικό για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της εφαρμογής καθώς και για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων να μπορούμε να τα συνδυάσουμε παραδείγματος χάρη. Οι δείκτες αυτοί που σας είπα είναι όλοι τέτοιοι ώστε όπου γίνεται μια παρέμβαση πρέπει τα κράτη-μέλη να τους χρησιμοποιούν και να μας αναφέρουν τους αριθμούς. Όλα αυτά στα πλαίσια ενός ευρύτερου πλαισίου που το λέμε performance framework και, όπου, το οποίο εξετάζουμε και παρακολουθούμε επί πολλά χρόνια. Αυτό το πλαίσιο θυμίζει στα κράτη-μέλη ότι το θέμα των δικτών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, να έχουμε δηλαδή ποιότητά τους των δικτών. Και επίσης ο σκοπός είναι να μην χαθούν πουθενά παρακολουθήσεις δαπανών. Να έχουμε δηλαδή μια σαφέστερη εικόνα ότι όποτε δεν είναι αποτελεσματική μια παρέμβαση να φανεί ποιο είναι το λάθος και αν χρειάζονται πρόσθετη πόρη. There are two, uh, dates in that... Υπάρχουν εδώ δύο βασικές χρονικές στιγμές. Η μία βρίσκεται στη μέση της προγραμματικής περίοδου όπου γίνεται αναθεώρηση του ενδιάμεσου αποτελέσματος του προγράμματος. Αυτό τα λέμε milestones γιατί βρίσκονται στο δρόμο προς την επίτευξη του τελικού στόχου που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος του προγράμματος. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι επίσημες ημερομηνίες αποτίμησης της εφαρμογής του προγράμματος. Έρχομαι τώρα στο επόμενο τμήμα της παρουσίασής μου που αφορά τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Οικονομική Διακυβέρνηση. Γιατί είναι σημαντική η σύνδεση αυτή, πρώτον, είναι ζωτικό να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε στην πολιτική συνοχή δεν υπονομεύεται από άλλη πολιτική σε κάποια χώρα ασταθή ή δεν αντιτίθεται στους στόχους που έχουμε συμφωνήσει με την πολιτική συνοχής. Δεύτερον, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να προσαρμόζονται τα προγράμματα για την περίπτωση που υπάρχουν απρόβλεπτες ε, κοινωνικές ή οικονομικές προκλήσεις. Ας πούμε μια ενεργειακή κρίση, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούν τα προγράμματα στην νέα αυτή κατάσταση. Η οικονομική διακυβέρνηση της πολιτικής σύνοχης μπορεί να περιγραφεί και με το τρίγωνο που βλέπετε εδώ. Από τη μία πλευρά υπάρχει η πολιτική συνοχή που παρέχει ή ενισχύει τις επενδύσεις. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα βέλος προς τα πάνω, πράγμα που δείχνει ότι χορηγούμε πόρους για τη χρηματοδότηση δαπανών υπέρ της ανάπτυξης. Και αυτό ιδίως σε περιόδους όπου ζητούν τα κράτη-μέλη αυστηρότητα δημοσιονομική και άρα η δημοσιονομική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά η πολιτική συνοχή επίσης συμβάλλει στην ενίσχυση δυνατοτήτων, οικοδόμηση δυνατοτήτων για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη και είπε και ο Νικόλας προηγουμένως ότι αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές και για μας στην πολιτική συνοχή. Υπάρχει μια σύνδεση λοιπόν και με τους όρους που θέτουν τα λειτουργικά προγράμματα ώστε οι επενδύσεις να μπαίνουν στο πλαίσιο, σε ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε τα κράτη-μέλη να προοδεύουν γενικότερα προς την επίτευξη του στόχου των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όλα αυτά συνδέονται στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εκασαμίνου. Αυτό το νέο πλαίσιο διασφαλίζει ότι συστάσεις αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα λαμβάνονται υπόψη και σε σύναψη εταιρικών συμφωνιών. Στην τωρινή φάση του προγραμματισμού των, προγραμμα... των σχεδίων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συστάσεις αναχώρα. Επίσης είναι φανερό ότι ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις θα είναι πραγματικά στοχευμένες και θα συνδέονται με τις υψηλότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ανάπτυξη και απασχόληση και προωθούν την συνοχή με, τις τα μακροοικονομικά προγράμματα και τη φορολογία. Μετά υπάρχει το θέμα της σύνδεσης αυτής μεταξύ μακροοικονομικής διακυβέρνησης και πολιτικής μας. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Ήδη υπήρχε το 2007-2013 σε εκείνη την προγραμματική περίοδο, αλλά ίσως λιγότερο δομημένο, <clears throat> λίγο πιο αδύνατο. Στη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές μεταξύ των αναχώρασης τάσεων και των παρεμβάσεών μας. Καλύπτει όλα τα ταμεία και σχετίζεται και με τους μηχανισμούς που εφαρμόζει, που έχει, που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξετάζει τη συμμόρφωση με τη διαδικασία διακυβέρνησης, δηλαδή ελλείμματα, μακροοικονομικές ανισορροπίες και οικονομικές προσαρμογές. Και ίσως επίσης γίνεται λίγο πιο αυτόματη, πιο αυτόματη σύνδεση από ό,τι στο παρελθόν με ορισμένα όρια που μπορεί να προκύπτουν από τις απαιτήσει του κάθε προγράμματος και που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάργηση ή σταμάτημα των πληρωμών ή και των δεσμεύσεων ακόμα. Στους μακροοικονομικούς όρους έχουμε δύο κατηγορίες, δύο, μία, δύο. Πρώτος, πιθανά αιτήματα αναπρογραμματισμού διαρθρωτικών ταμείων λόγω των αναχώρα συστάσεων. Δεύτερον, πιθανό πάγωμα της χρηματοδότησης αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν ό,τι πρέπει ή δεν εφαρμόζουν έναν από τους τρεις μηχανισμούς διακυβέρνησης που προβλέπουμε. Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε, κάναμε μια ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή του αναπρογραμματισμού και τα συμπεράσματά μας εκεί ήταν ότι θα χειριστούμε αυτόν τον αναπρογραμματισμό με μεγάλη φρόνηση και προσοχή. Καταλαβαίνετε ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικός, να είναι πολύ χρήσιμος, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, καθιστά πραγματική προσαρμογή και να μην διαταράσει την γενικότερη εφαρμογή και χρήση των κοντιλίων. Οι νέες αυτές διατάξεις είναι κάπως δοκιμαστικές γιατί το 2017 η Κομισιόν θα κάνει αναθεώρησή τους των μακροοικονομικών όρων δηλαδή και προβλέπεται εκεί να γραφτεί έκθεση και να συζητηθούν και τα ευρήματα, τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και αν χρειαστεί, προβλέπεται επίσης να προσαρμοστεί και το νομοθετικό υπόβαθρο και αν χρειαστεί η Κομισιόν θα αλλάξει πρόταση. Θα κάνει πρόταση προσαρμογών δηλαδή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ζωτικός και τον προσέχουμε ιδιαιτέρως. Γιατί προφανώς το Κοινοβούλιο πρέπει να πληροφορείτε εγκαίρως σε περίπτωση που χρειαστεί να εφαρμοστούν εξαιρέσεις ή να γίνει παρέμβαση για αλλαγή του προγράμματος και να αναλυφθεί κάποια δράση από την Κομισιόν και εμείς είμαστε αποδεσμευμένοι να σας πληροφορούμε εγκαίρως και εσείς μπορείτε να μας καλείτε για δομημένους διαλόγους. Επίσης είναι προφανές ότι αν αρθεί κάποια από αυτές τις ρήτρε, τότε η Κομισιόν επίσης θα πληροφορεί αμέσω το Κοινοβούλιο. Τώρα το τρίτο τμήμα της παρουσίασής μου. Τα δημοσιονομικά εργαλεία. Και αυτό από τα πολύ σημαντικά και πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη και το μακρινότερο λίγο μέλλον πέρα και από το 2020. Εκεί πρέπει να δούμε πώς να επενδύσουμε στην building capacity των χωρών μελών. Οι αριθμοί βέβαια που έχουμε είναι πολύ ασαφείς ε, και περίπου γιατί βασίζονται στα λειτουργικά προγράμματα όπως τα ξέρουμε σήμερα. 12 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για τα ή από μάλλον μέσω των δημοσιονομικών εργαλείων, δηλαδή περίπου το ίδιο ποσό με την προηγούμενη περίοδο 7 με 13. Αλλά το εύρος εφαρμογής τους στη νέα περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κεντρικά ενωσιακά εργαλεία όπως η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ που προβλέπει ότι η πολιτική συνοχή και χρήματα από αυτήν μπορούν να συνδυαστούν με χρήματα από το κόσμο και τον ορίζοντα 2020. Υπάρχει και η παραδοσιακή εναλλακτική λύση των ε, συγκεκριμένων μέτρων αναχώρα. Και υπάρχει και κάτι καινούριο σαν εκλογή και ευσύ δηλαδή off the self χρηματοδότηση, δηλαδή έτοιμα δημοσιονομικά εργαλεία που να είναι βέβαιο ότι συμφωνούν με τους κανόνες που εφαρμόζει κάποιο κράτος, να τα παίρνουν τα κράτη και να τα εφαρμόζουν όπως θέλουν γιατί είναι ασφαλή. Παρ' όλα αυτά τα δημοσιονομικά, στα δημοσιονομικά εργαλεία χρειάζεται περισσότερη τεχνογνωσία και γι' αυτό η Κομισιόν προσπαθεί να χορηγήσει τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη σε μία και μόνη δέσμη που την λέμε Φι Κόμπας και που έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται. Γιατί τονίζουμε τόσο πολύ τη χρήση αυτών των δημοσιονομικών εργαλείων, γιατί υπάρχει ένας πολύ σαφής λόγος. Όταν υπάρχουν σχέδια ή προγράμματα που αποφέρουν κέρδη, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δημοσιονομικά εργαλεία για να αντικαταστήσουμε υπάρχοντα ποσά. Έτσι θα γίνει πολύ μεγαλύτερη μόχυλευση. Επίσης, στη νέα προγραμματική περίοδο δεν έχουμε θεματικούς περιορισμούς. Είναι ορθάνυχτη στην εφαρμογή οποιοδήποτε δημοσιονομικού εργαλείου της ταιριάζει περισσότερο. Με βάση μόνο το κριτήριο να αποφέρουν κέρδος στα προγράμματα. Ιδιαίτερα τονίσαμε τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο παρελθόν. Η ΜΜΕ ήταν ο κύριος ωφελούμενος από τέτοια προγράμματα και το ίδιο θα γίνει μάλλον και στο μέλλον. Και η πρωτοβουλία των ΜΜΕ θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στήριξής τους. Μέχρι τώρα δύο χώρες έχουν ζητήσει τέτοια στήριξη, Ισπανία και Μάλτα. Και μερικές ακόμα το σκέφτονται. Η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ελλάδα. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι τα δημοσιονομικά αυτά εργαλεία σχετίζονται με τη γενική πολιτική και προγράμματα της Ένωσης. Αυτό αποσαφηνίστηκε στα προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου Γιούνκερ να είμαστε πιο φιλόδοξοι και για την πολιτική συνοχή για συνεργασία με τα δημοσιονομικά εργαλεία. Έχουμε περίπου το ίδιο επίπεδο που ζήτησαν τα κράτη-μέλη και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να έχουμε σαν στόχο σχεδόν τον διπλασιασμό των δημοσιονομικών εργαλείων που χορηγούμε για την περίοδο 14 με 20 αντί να συνεχίσουμε απλώς όπως την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομερέστατη αυτή παρουσίαση. Πριν από δύο εβδομάδες συζητήσαμε και εμείς εδώ τους όρους, τους μακροοικονομικούς όρους και ήταν πολύ πολύ πλοκή μακρά η συζήτηση, αλλά είμαι βέβαιη ότι και σήμερα υπάρχουν απορίες. Ορίστε κύριε Άντριτσμό. Ευχαριστώ. Άλλη μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τώρα, μα είπατε πώς μπορείτε να σταματήσετε τη χρηματοδότηση για κάτι, ενώ θεωρητικά. Ένα έργο είναι στη μέση, παραβιάζουν τους κανόνες ε, και πρέπει να σταματήσει. Ή πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή εάν η χώρα δεν συμφωνεί με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και έχει άλλες προτεραιότητες. Θα πείτε όχι σε όλη τη χρηματοδότηση αυτής της χώρας. Ακόμα και αν είναι καθαρός φορέας, γιατί τα δικά του λεφτά ανακυκλώνονται με τις δικές σας προτεραιότητες. Ευχαριστώ κύριε Έθεριτς. Κυρία Βάνα, εγώ μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω. Μπορείτε να αναφερθείτε στην ρήτρα επενδύσεων που αναφέρθηκε από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Γιατί υπόθηκε ότι θα μπορούσαν να βγουν οι επενδύσεις έξω από το κριτήριο του ελλείμματος. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Απαντήστε λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Με συγχωρείτε, ε, δεν είμαι σίγουρος για την ερώτηση του κυρίου. Κοιτάξτε, ε, το πρώτο ήταν έστω ότι έχει, έχουμε ένα σχέδιο που έχει γίνει το μισό και μετά δεν είναι σε γραμμέ. γραμμές. Τι, τι γίνεται. Δεύτερον, αν μια χώρα δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες και έχει άλλες προτεραιότητες. Κόβεται όλες τις αιτήσει. Ακόμα και σε περίπτωση καθαρού εισφορέα ανακυκλώνετε τα δικά τους χρήματα με τις δικές σας προτεραιότητες. Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ναι, μάλιστα. Στο πρώτο μιλάτε για επίπεδο έργου και κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ποιες κατευθυντήριες γραμμές λέτε. Γιατί εμείς μιλάμε για την πολιτική συνοχής. Στο πλαίσιο δηλαδή των προγραμμάτων αυτών μιλάμε. Έχουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα που έχει υιοθετηθεί από την Κομισιόν που παρουσιάζει βασικές προτεραιότητες ε, δαπανών, ξέρω εγώ, έρευνα και καινοτομία με τρεις άξονες προτεραιότητας που λένε ποιοι είναι οι στόχοι, πώς θα επιτευχθούν και τους στίχους των τίτλων. Είναι μετά, αρχή, είναι μετά δουλειά της διαχειριστικής αρχής να επιλέξει τα έργα. Η Κομισιόν δεν κοιτάει το κάθε έργο. Αυτό το κάνει το καράτος μέλος. Οπότε προφανώς θα συμμορφώνεται με τους κανόνες επιλεξιμότητας και θα πετυχαίνει αυτούς τους στόχους. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι να έχει κακές επιλογές σε όλα τα έργα και δεν έχει άρα τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. και μετά όταν θα έρθουμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, αν δεν έχετε βεβαίως ε, επιτύχει τα αποτελέσματα, θα υπάρξει μια διόρθωση. Όχι λόγω μεμονωμένου έργου, αλλά γιατί δεν έχετε επιτύχει ε, τους γενικούς στόχους. Για το δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή σιωθετηθεί ε, το πρόγραμμα από την ε, Κομισιόν δεν μπορούμε να πούμε μετά όχι αλλάξαμε γνώμη, δεν μας αρέσει. Ε, δηλαδή υπάρχει μια βεβαιότητα έτσι και μια σταθερότητα. Και υπάρχει μετά η διαβεβαίωση ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Η μόνη δηλαδή πραγματική εξουσία που έχει η Κομισιόν για να επιβάλλει αλλαγή στις δαπάνες είναι μέσω αυτού του όρου που αφορά τις ε, συστάσεις χώρα. Αν έχει συμβεί δηλαδή κάτι σοβαρό και το Συμβούλιο κάνει μια σύσταση ε, και λέει, ξέρω εγώ, θα πάτε τα λεφτά σας εκεί. Δηλαδή αυτά τα σενάρια που λέτε δεν μπορούν να συμβούν κανονικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τη ρήτρα επενδύσεων, πιστεύω και από γνωρίζω, αυτό που ελέγχθη πρόσφατα ε, με βάση την παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου σχετίζεται με ένα νέο μέσο που προτάθηκε να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις παρά το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο. Όπως ξέρετε, στην περίπτωση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων υπήρξε ένα ελάχιστο περιθώριο ευελιξίας αναπερίπτωση στο παρελθόν, αλλά όπως γνωρίζουμε, οι κανόνες του παιχνιδιού δεν θα πρέπει να επανεξεταστούν σε αυτή τη φάση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση σχετίζεται με ενδεχόμενες συνεισφορές των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια του νέου μέσου που θα δημιουργηθεί. Ε, δεν σχετίζεται άμεσα με τη δική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίσλερ. Και τώρα συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος της ε, ε, συνεδρίασης. Ο κύριος Φρανκ Σεμπέρτ έχει το λόγο, ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για θέματα διαχείρισης και ελέγχου. Έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Θα στραφώ τώρα σε θέματα πρακτικής εφαρμογής, έμπρακτης εφαρμογής. Είναι μια πολύ καλή εισαγωγή αυτή που μας έδωσε ο Νίκολας. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ορισμένα λόγια για τα εθνικά συστήματα ελέγχου και τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών σε σχέση με την ε, καθημερινή εφαρμογή των προγραμμάτων. Μετά θα μιλήσω για τις ε, ευθύνες ελέγχου που επιμερίζονται μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής και θα μιλήσω και για τα διάφορα μέσα για την νομιμότητα και την τακτικότητα των ε, χρηματοδοτήσεων εκεί όπου υπάρχουν αναστολές και αναβολές καθώς και οι χρηματοοικονομικές διορθώσεις που ισχύουν για τη νέα περίοδο. Θα αρχίσω με αυτή την πυραμίδα για να σας δείξω ποια είναι αυτά τα μπλοκ διασφάλισης για τα προϊόντα αυτά και για την νομιμότητα και τακτικότητα της ε, χρηματοδότησης. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο γεγονός, όπως βλέπετε στην δεξιά πλευρά της γραφικής παράστασης, ότι έχετε στοιχεία πριν από την έγκριση των προγραμμάτων, οι διαπραγματεύσεις, η διαδικασία διορισμού και εγγυήσεων σε σχέση με την τακτικότητα των μελλοντικών δαπανών και έχετε και τις δράσεις ή προαπαιτούμενα κατά την εφαρμογή από πλευράς διαχείρισης, πιστοποίησης, ελέγχων μέχρι την, τον έλεγχο της Επιτροπής. Βλέπετε ότι υπάρχει επιμερισμένη ευθύνη μεταξύ των ε, κρατών μελών, των τριών αρχών δηλαδή ως προς τη διαχείριση, πιστοποίηση ή έλεγχο και ο ρόλος της Επιτροπής για την επίβλεψη. Μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινή διαχείρισης και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο στα πλαίσια αυτού του επιμερισμού. Και έτσι έχουμε μία σειρά γενικών αρχών που θα πρέπει να τηρηθούν από όλα τα συστήματα ελέγχου, ιδιαίτερα την περιγραφή των λειτουργιών από τις διάφορες αρχές, διαφορά λειτουργιών σε σχέση με την τακτικότητα, τον τακτικό χαρακτήρα των δαπανών καθώς και μηχανογραφημένα συστήματα ελέγχου και λογοδοσίας. Και ένα σύστημα για τον έλεγχο και επιστοποίηση όλων των συστημάτων. Τέλος, συμφωνίες ελέγχου για όλα τα προγράμματα έτσι ώστε να υπάρξει η ανείχνευση και η διόρθωση όλων των παρατυπιών και απάτης. Η λέξη απάτη προσετέθη στον κανονισμό για την περίοδο 14 με 20. Πώς, ε, έχει, λοιπόν, πώς έχουν οι λειτουργίες της διαχειριστικής αρχής. Υπάρχει μια διαχειριστική αρχή η οποία θα πρέπει να σταθεί στις αρχές της ε, χρηστής ε, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και όπως είπε και ο Νίκολας, ε, καταρχήν επιλέγουν τα προγράμματα που σχετίζονται με τα κριτήρια και τις προτεραιότητες του προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι, όλα αυτά τα προγράμματα εντάσσονται στους στόχους και στις προτεραιότητες, να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι για την νομιμότητα και τακτικότητα των χρηματοδοτήσεων και οι δικαιούχοι, δημόσιοι ιδιωτικοί φορείς θα εφαρμόσουν την πολιτική ή το project, αλλά οι δικαιούχοι θα πρέπει να κατανοήσουν πολύ καλά το ρόλο τους και τις ε, υποχρεώσεις τους με βάση τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος, ε, δηλαδή πώς θα πρέπει να τηρήσουν τους διάφορους νόμους ε, κατά την λογοδοσία στις διάφορες αρχές με βάση και τα τελικά προγράμματα ή υπηρεσίες και με βάση τις αρχές της διαχειριστικής αρχής. Αυτό έχει σημασία για την επιλεξιμότητα των ε, σχεδίων και θα πρέπει να ε, συμμορφώνονται με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής αρχής. Επίσης θα πρέπει ο δικαιούχος να μπορέσει να ε, εφαρμόσει αυτά τα σχέδια και θα πρέπει να γίνονται επαληθεύσεις, διαχειριστικές επαληθεύσεις για επιστροφή χρημάτων έτσι ώστε οι δαπάνες συμβαδίζουν με την πρόοδο των προγραμμάτων που εφαρμόζονται επιτοπίως. Και αυτές οι επαληθεύσεις είναι και το πρώτο χαράκομα κατά των ε, παρατυπιών γιατί δεν πιστοποιούνται οι δαπάνες εάν υπάρχουν προβλήματα στη δήλωση δαπανών. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να το κάνει αυτό μέσω διοικητικών ελέγχων ε, έτσι ώστε να υπάρχει λογοδοσία μέχρι και το τελευταίο ευρώ δαπανών με απλές τεχνικές με έγγραφα υποστήριξης για την επιλεξιμότητα της δαπάνης και θα πρέπει να γίνονται και επιτόπιες έρευνες έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι και να γίνονται επαληθεύσεις ότι δηλαδή όλες οι δηλώσεις συμβαδίσουν με τις δηλώσεις λογοδοσίας. οι ίδιες διατάξεις που είχαμε και την περίοδο 2007-2013 για τις επαληθεύσεις έχουμε και τις, ε, τους ετήσιους λογαριασμούς. Η διαχειριστική αρχή λοιπόν θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι μέχρι ότου πιστοποίηση τους λογαριασμούς όλοι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται για να ανοιχνευθούν παρατυπίες και να απορριφθούν σχέδια. Υπάρχουν όμως και νέες απαιτήσει. Θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα κατά της απάτης. Σας είπα ότι αυτή η τυπολογία των παρατυπιών και η λέξη απάτη που εισήχθη στον κανονισμό ορίζει τα μέτρα κατά της απάτης που εντάσσονται στο σύστημα πέρα από τον έλεγχο του κανονισμού. Αυτά τα μέτρα κατά, τον, κατά της απάτης θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά να καταπολεμηθεί η απάτη, αλλά θα πρέπει να είναι αναλλαγικά και ως προς τον κίνδυνο. Δηλαδή, μερικά προγράμματα ε, προβλέπουν πολύ λίγα επιπρόσθετα μέτρα διότι τα συστήματα έχουν τη σχετική στεγανοποίηση κατά της απάτης. Υπάρχει και το μέσο αποτίμησης κινδύνου που προβλέπει η Επιτροπή. Επιτροπή. Για την καταπολέμηση της απάτης. Από πλευράς διαχειριστικής αρχής και της λογοδοσίας της υπάρχουν δύο προαπαιτήσεις θα πρέπει να υπάρχει μία δήλωση διαχείριση που αποστέλλεται στην Επιτροπή κάθε χρόνο με βάση τη λειτουργία του συστήματος και για τη νομιμότητα και τακτικότητα των πληρωμών. Αυτό έχει σημασία γιατί αποτελεί δέσμευση της διαχειριστικής αρχής ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες της και προβαίνει σε όλες τις δράσεις έτσι ώστε να υπάρχει τακτικότητα, νομιμότητα και καταπολέμηση της απάτης και, το, και οι σωστοί δείκτες εκρών. Παράλληλα, αυτή η δήλωση διαχείρισης θα πρέπει να συνοδεύεται και από, ένα, από μια ετήσια σύνοψη για τους ελέγχους, ε, τα project που αναγνωρίζουμε και να αναφερθεί στην Επιτροπή ποιο είναι το follow-up όλων των ε, εκθέσεων ελέγχου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο μέσα στα πλαίσια του πακέτου αυτών των εγγράφων. Αυτά για τη διαχειριστική αρχή που είναι ο πυλώνας εφαρμογής των προγραμμάτων. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή πιστοποίησης. Γιατί πιστοποίησης, γιατί αυτή η αρχή θα πρέπει να πιστοποιήσει τις δαπάνες στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και είναι υπεύθυνη για την καταβολή πληρωμών στους ε, δικαιούχους. Η αρχή αυτή θα πρέπει να υποβάλει ε, δηλώσεις, μάλλον αιτήσει πληρωμών στην Επιτροπή από την 1η Ιουλίου μέχρι την ε, μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και οι δαπάνες να βασίζονται σε αξιόπιστα συστήματα λογαριασμών, σχετικά έγγραφα και επαληθεύσεις. Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να έχει ένα σύστημα πληροφορικής όπου να πιστοποιεί κάθε πράξη ως προς τις ενδεχόμενες διορθώσεις και ούτω καθεξής. Και αυτό το νέο στοιχείο για την περίοδο 14-20. Η αρχή πιστοποίησης συμπληρώνει τους λογαριασμούς στο, έ, τέλος του έτους και πρέπει να αποστείλει αυτούς τους λογαριασμούς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για πλήρη έγγραφα και η αρχή πιστοποίησης θα παληθεύσει αυτούς τους λογαριασμούς που θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια της ε, νομιμότητας και τακτικότητας πληρωμών με όλους τους ελέγχους που γίνονται για το πρόγραμμα αυτό. Επίσης προβλέπει ότι η αρχή πιστοποίησης ίσως συγχωνευτεί με την διαχειριστική αρχή, ανάλογα με τις ανάγκες. Η τρίτη αρχή για κάθε πρόγραμμα είναι η ελεγκτική αρχή. Για την περίοδο 7-13 η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να ορίσει μία τακτική και στρατηγική ελέγχου για ολόκληρη την περίοδο και αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην Επιτροπή αν ζητηθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι ίσως ε, μέσα στα πλαίσια του κανονισμού η διαχειριστική και αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να οριστούν από τα κράτη-μέλη αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα εξάρτητο, μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου με βάση κριτήρια ως προς τις ε, κοινέ προδιαγραφές. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε πληροφορίες, δηλαδή ότι θα υπάρχει αυτό το ανεξάρτητο σώμα ή αρχή μέσα στα πλαίσια της έγκρισης των προγραμμάτων. Τη στιγμή που έχει οριστεί η ελεγκτική στρατηγική κατά την περίοδο εφαρμογής γίνονται έλεγχοι την πραγματική λειτουργία των συστημάτων με όλα τα προαπαιτούμενα του κανονισμού. και υπάρχουν 18 όροι που πρέπει να πληρούνται σε όλα τα προγράμματα. Και επίσης η Επιτροπή θα ελέγξει το κατά πόσο πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Επίσης, περιλαμβάνει θεματικούς ελέγχους σε σχέση με την αξιοπιστία δικτών εκρών για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και σχετίζεται με τομείς υψηλού κινδύνου ως προς την επαλήθευση και έλεγχο διαδικασιών διαγωνισμού ή την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της απάτης. Και αυτό γίνεται χρόνο με το χρόνο με το follow-up της αρχής. Επίσης κάθε χρόνο θα πρέπει να διενεργήσει ελέγχους με βάση συγκεκριμένα ε, δείγματα, αντιπροσωπευτικά δείγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφανθούμε για την λειτουργία του συστήματος. Τα δείγματα αυτά των πράξεων σχετίζονται με δαπάνες για τη χρήση από τον Ιούλιο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο και επίσης θα πρέπει να ε, διενεργούνται έλεγχοι επί των λογαριασμών στοιχεία που επιβάλλονται στην Επιτροπή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Αυτή η εργασία επιβαρύνει την ελεγκτική αρχή από το 16 και μετά, έτσι ώστε να παρέχει στην Επιτροπή ένα ε, έλεγχο, μία έκθεση μάλλον σε σχέση με την ομότητα και την τακτικότητα αυτών των πληρωμών και την ε, ουσιαστική λειτουργία του συστήματος κατά την χρήση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προβεί σε μια εποπτεία και με βάση προγράμματα που υπερβαίνουν τα 250 εκατομμύρια η Επιτροπή θα πρέπει να ε, ε, μπορεί μάλλον να ζητήσει την επαλήθευση του πακέτου. Εκεί που έχει ε, αναλάβει, στο έργο που έχει αναλάβει, προβαίνει σε προληπτικούς ελέγχους. Συνεργαζόμαστε με τις ελεγκτικές αρχές για να τους δώσουμε στοιχεία, μεθοδολογικά μέσα, ε, καταλόγους ελέγχου και ούτω καθεξής. Και οι, οι, οι αρχές αυτές θα πρέπει να συνεργαστούν ως προς το ΕΚΤ, ΕΤΠΑ κλπ. Έχουμε μία ενιαία ελεγκτική στρατηγική για το 14-20 με μέτρα για τον έλεγχο, εκεί που είναι αναγκαίο. Επίσης υπάρχει συντονισμός με τις ελεγκτικές αρχές, ε, σκεφτόμαστε κάθε χρόνο για να γίνονται έλεγχοι και να, για να έχουμε μία ενιαία διαδικασία ελέγχου και για μείωση του όγκου του ελέγχου όταν μπορούμε να βασιστούμε στις εθνικές ελεγκτικές αρχές για να έχουμε αναλογικό έλεγχο και για να μειώσουμε τον όγκο ελέγχου των δικαιούχων. Η εργασία ελέγχου από την Επιτροπή κάθε χρόνο ασχολείται με αυτές τις δηλώσεις αξιοπιστίας που θα πρέπει να λάβουμε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου έτσι ώστε να φτάσουμε σε συμπεράσματα για την αποδοχή των λογαριασμών, την αξιοπιστία, τη δήλωση αξιοπιστίας και τις δαπάνες δυνάμει των λογαριασμών και για να φτάσουμε σε στοχοθετημένους ελέγχους σε προγράμματα όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την, τις παρατυπίες. Με βάση τους ελέγχους συμμόρφωσης η Επιτροπή ίσως θα πρέπει να προωθήσει μια διαδικασία χρηματοοικονομικών διορθώσεων και υπάρχουν ορισμένοι όροι που ορίζονται από τον κονισμό για να γίνουν διορθώσεις. Για να φτάσει στην δήλωση ναι. αξιοπιστίας, η Επιτροπή έχει μία σειρά μέσων για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Η διακοπή πληρωμών είναι μια ε, γνωστή διαδικασία, πρόκειται για έξι μήνες, εκεί όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ελλείψεις στα προγράμματα και όπου η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε επιπρόσθετους ελέγχους για παρατυπίες. Υπάρχει και ένας νέος όρος που ορίζεται για την περίοδο 14-20, εκεί όπου τα κράτη-μέλη δεν στείλουν μία από τις πέντε δηλώσεις αξιοπιστίας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα γιατί και αυτό το μέσο είναι το ίδιο. Αυτό αφορά και τις αναστολές πληρωμών. Εδώ η Επιτροπή μπορεί να σταματήσει, να, ε, σταματήσει τις ενδιάμεσες πληρωμής τη στιγμή που υπάρχουν υπάρχουν στοιχεία για ελλείψη στη διαχείριση ή στη δήλωση πληρωμών. Επίσης, ε, μπορεί να γίνει αναστολή πληρωμών όταν το κράτος μέλος δεν έχει επιλύσει τις ε, καταστάσεις. Υπάρχουν όμως και νέοι όροι, στους οποίους αναφέρθηκε ο Ρούντολφ. Ρούντολφ σε σχέση με ζητήματα χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Αυτό που ε, είναι ένα νέο στοιχείο είναι το τρίτο μέσο που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της. Δηλαδή η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει καθαρές χρηματονομικές διορθώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει από τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια τις ε, επιμερισμένες διαχειρίσεις τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διορθώσουν αυτές τις παρατυπίες. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγξουν όλες τις πράξεις, τις σχετικές πράξεις που σχετίζονται με αυτή την παρατυπία. Όταν το κράτος ε, μέλος ε, ανοιχνεύσει μία παρατυπία και προβεί στις οι οικονομικές διορθώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ποσά αυτά για άλλες ε, πράξεις που είναι επιλέξιμες. Έτσι, τα κράτη-μέλη έχουν κίνητρα για την έγκαιρη διαδικασία ελέγχου η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει ελέγχους και διορθώσει όταν υπάρχουν πολλές ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων που δεν έχουν διορθωθεί από τα κράτη-μέλη. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας ε, των διορθώσεων, το καινοτόμο στοιχείο και το νέο νομικό μέσο που διαθέτει η Επιτροπή στο ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο ναι. είναι να προβεί σε καθαρές οικονομικές διορθώσεις αν η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανοιχνεύσει παρατυπίες στην πραγματική λειτουργία των συστημάτων μετά από την υποβολή των λογαριασμών και της δήλωσης αξιοπιστίας. Υπάρχουν όροι που αφορούν την έλλειψη δήλωσης ε, παρατυπιών προγενέστερα από το κράτος μέλος. Αυτές οι διορθώσεις θα πρέπει να βασίζονται στις ε, παρατυπίες οι οποίες έχουν ανοιχνευθεί, αλλά όταν η παρατυπία ή η έλλειψη είναι συστημική, τότε θα πρέπει να γίνονται όχι μόνο με μονομένες διορθώσεις, αλλά να ποσοστοποιηθεί σε ένα καταποκοπή ποσό η αποκατάσταση της παρατυπίας ε, που ε, αφορά ένα φάσμα από 5 μέχρι 100%. Αυτά τα καταποκοπή ποσά αφορούν τις συνολικές ε, δαπάνες. εκεί που εφαρμόζονται τα καταποκοπή ποσά ανεξάρτητα από τις πράξεις. Όταν δεν είναι αναλογικά αυτά τα μέτρα υπάρχει δυνατότητα μείωσης αλλά εκεί όπου υπάρχουν παραβιάσεις, oh. συνεχείς παραβιάσεις μπορεί να αυξηθούν τα ποσά, αυτά τα καταποκοπήν ποσά στον ανώτατο, στο ανώτατο όριο. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την νομιμότητα και τακτικότητα των πληρωμών και για να υπάρχουν κατάλληλες εγγύσεις προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ερωτήσει μετά από όλα αυτά. σύντομη γιατί ήσασταν πολύ αναλυτικός. Αλλά αν το είπατε ζητώ συγγνώμη. Αλλά ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ελεγκτών σε ένα κράτος μέλος. Πρέπει να είναι οροκοτή, ε, κάποια πιστοποίηση όπως έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναχώρα, πώς πάει το σύστημα. Μάλιστα, άλλες ερωτήσεις. Πράγματι. Αναλυτική η παρουσίαση. Να αναφερθώ τώρα σε αυτά που ψηφίσαμε πριν καταπολέμηση της απάτης. Οι περισσότεροι εδώ μέσα θεωρούσαν πως πρέπει να αντιμετωπιστεί απάτη, αλλά υπάρχει ανησυχία. Πώς ε, υπάρχουν κάποιες παρατυπίες που οφείλονται μόνο και μόνο στην πολυπλοκότητα του ε, συστήματος. Εσείς θεωρείτε πως οι κανονισμοί αυτοί όπως τροποποιήθηκαν είναι βελτίωση. Όταν λέω βελτίωση όμως εννοώ μόνο απλοποίηση και αποτελεσματικότητα, όχι περισσότερους ελέγχους. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μπορείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις αρχές του δημοσιονομικού ελέγχου. Δεν χρειάζονται πιστοποίηση από την Κομισιόν. Ορίζονται από τα κράτη-μέλη, ιδίως από τα Υπουργεία Οικονομικών τους. που έχουν τέτοιες υπηρεσίες. Συνήθως πρόκειται για επαγγελματίες, πρέπει να εργάζονται ανάλογα με τα διεθνή ελεγχτικά πρότυπα και το κράτος πρέπει να επιτηρεί. Κατά την περίοδο 7 με 13 έγιναν 47 έλεγχοι των αρχών και καταλήξαμε ότι 43 από αυτές τις αρχές είναι αξιόπιστες και εργάζονται με βάση όλα τα δέοντα κριτήρια. Ακόμη και αν λοιπόν δεν υπάρχει επίσημο πλαίσιο ορισμού, καθορισμού αυτών των αρχών, σας διαβεβαιώνω ότι συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες που σέβονται διεθνή πρότυπα. ώστε να επεξεργαστούμε μαζί τη μεθοδολογία και τα κριτήρια των ελέγχων. Μερικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα βέβαια. Αυτό εξαρτάται από τη διοικητική τους δομή, αλλά οι αρχές του δημοσιονομικού ελέγχου είναι πάντοτε ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Αλλιώς ζητούμε διόρθωση. Σε μερικές περιπτώσεις δεν ήταν τέτοιοι. Εγώ θα επανέλθω στη δεύτερη ερώτηση. Όπως είπε και ο Φραγκ, το βασικό στοιχείο είναι ότι πρέπει να σέβονται τους τα διεθνή πρότυπα δημοσιονομικών ελέγχων. Το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Λόα επανέρχεται σε αυτό το θέμα της απλοποίησης. Δεν είναι τόσο η δημοσιονομική έλεγχη, αλλά οι κανόνες μάλλον που πρέπει να εφαρμόζονται για να εγκριθεί και να θεωρηθεί νομότυπη δαπάνη. Όπως είπατε και εσείς βέβαια περισσότεροι κανόνες σημαίνουν και περισσότερες ατασταλίες ίσως αλλά ένας από τους στόχους στο νέο κανονισμό ήταν ακριβώς η απλοποίηση. Υπάρχουν τρόποι για να επιτευχθεί αυτό μέσω της μείωσης ορισμένων κριτηρίων ε, έγκρισης και απλοποίησης κόστους Ας πούμε ένα κράτος μέλος μπορεί να πει θα χρησιμοποιήσουμε το στάνταρ κόστος αντί να χρειάζεται δηλαδή να δικαιολογήσουμε το κάθε ευρώ να χρησιμοποιούμε έναν προβλεπόμενο έτοιμο τρόπο. Να μην χρειάζεται οι αρχές που κάνουν τον έλεγχο να υποβάλουν το κάθε εισιτήριο λεωφορείου που χρησιμοποιούν κτλ. Μερικά βέβαια δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Το Περιφερειακό Ταμείο χρησιμοποιεί δημόσιες προσφορές και προμήθειες και γι' αυτό ισχύουν οι σχετικές οδηγίες και πρέπει να εφαρμόζονται αυτές. Αν διαβάσετε την έκθεση, την ετήσια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, βλέπετε ότι στον τομέα μας Πολλά από τα λάθη που βρίσκουν σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες. Αλλά από αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε γιατί ε, είναι ο προβλεπόμενος ο νομισμένος τρόπος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, να τους δώσουμε οδηγίες. Απλοποίηση λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα κράτη-μέλη κάνουν τους κανόνες ε, έγκρισης των προγραμμάτων και εμείς παρακολουθούμε, επιτηρούμε πολύ στενά τι συμβαίνει. Έτσι μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν υπερβολικά πολλοί κανόνες που οδηγούν σε περισσότερα λάθη. Ευχαριστούμε πολύ κύριοι για τις παρουσιάσεις σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και άλλα ερωτήματα στο μέλλον. Αλλά περιμένετε υπομονή. Επόμενο σημείο μας είναι τα διάφορα. Δεν βλέπω να υπάρχουν διάφορα. Τελειώνει η συνεδρίασή μας εδώ. Η επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 3 με 6,5 εν Βρυξέλλες και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 9 με 12,5 με 12,5 ευχαριστώ τις διερμηνεύτριες και κλείνει εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής Περίφ για σήμερα.